Colleagues, uh, please take your seats. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Can you please uh, close the doors and please take your seats. Καθίστε παρακαλώ και κλείστε την πόρτα για να αρχίσουμε. Okay, please take your seats immediately. It's a hearing. all members your seats? Πρέπει να αρχίσουμε την ακρόαση. Καλησπέρα σας. Είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια σήμερα και ήδη έχουμε δυστυχώς ε, καθυστερήσει ε, κάποια λεπτά. Ε, οπότε θα περάσω απευθείας στην ακρόαση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω να, σας καλωσορίσω όλους, να καλωσορίσω εξ ονόματος όλων ε, την ε, κυρία Ραϊχέρτς, ε, τους συναδελφούς από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και των Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Δύο φίλων και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην επιστολή της 3ης Ιουλίου ο πρόεδρος Μπαρόσο ανέφερε ότι αν διοριστεί η Επίτροπος θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, η θαγένεια. Ε, μόλις ολοκληρώσω ο νέο πρόεδρος, ο κύριος Φόποτα και η κυρία Καρσία Περές που είναι πρόεδρος Επιτροπής ε, Γυναικών θα πάρουν το λόγο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την αρχική δήλωση της κυρίας Ρέιχελτς. Στη συνέχεια μόνο οι συντονιστές θα πάρουν το λόγο βάσει των συμπεφωνημένων ανάμεσα στους τρεις προέδρους η, όπως αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων, η ακρόαση δεν θα υπερβεί τα 90 λεπτά. Ε, και μέσα σε αυτά τα χρονικά περιθώρια θα οργανώσουμε τις ερωταπαντήσεις και ξαναλέω θα παρεύουν μόνο οι συντονιστές. Ε, θα ήθελα να στήσω συγγνώμη τα υπόλοιπα μέλη ε, των Επιτροπών αλλά λόγω της έκτακτης φύσης αυτής της ακρόασης για το αξίωμα περιορισμένης διάρκειας θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Οι κανονικές ακροάσεις θα γίνουν το φθινόπωρο. Έχετε διαδικαστικό, μπορείτε να μας πείτε ποια είστε Σα eh, eh. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Μάιερ, Βίκη Μάιερ είναι το όνομά μου. Είμαι του κόμματος της Ελευθερίας μέλος. Ακόμα είμαι μη εγγεγραμμένη. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραπονέθηκα για το ότι δεν μπορώ να διατυπώσω ερώτηση. Και αυτό το παράπονο θέλω να το υπογραμμίσω εδώ. Εμείς οι μη εγγεγραμμένοι πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να λάβουμε τον λόγο και να παρέμβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που προβάλλατε με αποτελεσματικό και ευγενικό τρόπο την ένστασή σας. Ε, τη σημειώνουμε και θα περάσουμε ε, στις δηλώσεις του κ. Σφόποτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, Πολιτικών Ελευθεριών, και δικαιωμάτων των γυναικών αυτών των κοινοβουλευτικών επιτροπών αλλά επίσης πρώτα και την κυρία Μαρτίν Ράιχερτς την υποψήφια επίτροπο Θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών μας επιτροπών είναι πολύ σημαντική υπόθεση επειδή υπάρχουν τομείς ε, μέρη κοινού ενδιαφέροντος ε, για μας από κοινού όλους επίσης τομείς ευθύνης από την ίδια την υποψήφια επίτροπο που επικαλύπτονται με τα πεδία αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για παράδειγμα ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική δικαιοσύνη και το οικογενειακό δίκαιο και το <clears throat> ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Αυτή είναι η τομή όπου τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων σε αυτά τα θέματα θα επικεντρωθούν στις ερωτήσεις τους. Κυρία, βέβαιος ότι μετά την εκλογή σας η συνεργασία μαζί σας θα είναι πολύ γόνιμη. Τόσο γόνιμη όσο ήταν και κατά το παρελθόν με την ίδια την κυρία Επίτροπο, κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ, όταν ήταν εκείνη η Επίτροπος. Μια και πιέζει ο χρόνος, ας δώσω τον λόγο στη συνέχεια στην κυρία Γκαρσία Πέρες, παρακαλώ, από την Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και στις συναδέλφους. Καλώς ήρθατε κυρία Ράιχερτ. Από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας παίρνω το λόγο και θέλω να πω ότι θεωρούμε ότι η αρμοδιότητά σας είναι σημαντική. Έχετε το καθήκον στην περίοδο κατά την οποία ε, θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας ε, να ε, συνεχίσετε την πολιτική ισότητας και γι' αυτό θα σας ρωτήσουμε σε αυτή τη συνεδρία. Η πολιτική για την ισότητα θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Μιλούμε για την καταπολέμηση της βίας ε, στα φύλλα, στα δύο φύλλα. Μιλούμε για τις άδειε μητρότητα, μιλούμε για την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Μιλούμε για την κατάσταση ε, που βιώνουν οι γυναίκες σε περίοδους κρίσης για τα δικαιώματα στην αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία. Όλα αυτά τα θέματα είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή για τις, γυναίκες, για τις γυναίκες και θα σας τεθούν από τις διάφορες συντονίστριες κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασης. Ας περάσουμε ε, στις παρεμβάσεις από τους συναδέλφους από πλευράς Επιτροπών. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστούμε η Ράτσι. Θα ακούσουμε τις αρχικές δηλώσεις της κυρίας Ρέιχαρτς. Φυσικά για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών το χαρτοφυλάκιό σας έχει ιδιαίτερη σημασία, οπότε έχετε στη διάθεσή σας ένα δεκάλεπτο για τις αρχικές σας δηλώσεις. Παρακαλώ. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να μιλήσω γαλλικά, εάν ε, μου επιτρέπετε, διότι μου δώσ, ε, σπούδασα νομικά ε, στα γαλλικά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ήθελα να προετοιμάσω ψυχολογικά τους διερμηνείς. Η παρουσία μου σήμερα εδώ απορρέει από την εκλογή της κυρίας Ρέντιν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να τη συγχαρώ. Από τη μία πλευρά η δική μου θητεία θα είναι εξαιρετικά σύντομη γιατί θα διαρκέσει μέχρι τη σύσταση σε σώμα της νέας Επιτροπής. Ωστόσο το γεγονός ότι μια Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζεται υποψήφια για τη θέση του Επιτρόπου είναι μια πρόκληση και μια ευθύνη για μένα και γνωρίζω το πόσο σημαντικό είναι. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιαστώ εδώ με κάθε δυνατή μετριοπάθεια. Θέλω να συνεχίσω τη δράση της κυρίας Ρέντιν τα τελευταία πέντε χρόνια και θα ήθελα να συνεχίσω και τη δική μου δουλειά μέχρι σήμερα, ε, να εξυπηρετήσω το γενικότερο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό άλλωστε είναι το κίνητρο που καθοδηγεί τις πράξεις μου καθημερινά τα τελευταία 30 χρόνια. Στις απαντήσεις στις γραπτές που έδωσα στο ρηγματολόγιο ε, πιστεύω ότι κατάφερα να αναπτύξω ε, τις θέσεις μου. Εάν τελικά οριστώ επί Επίτροπος, θα ήθελα να δηλώσω ότι θα συμμετάσχω πλήρως ε, με φιλική, με συναδελφική ατμόσφαιρα, με πνεύμα συνεργασίας αλλά και με πλήρη ανεξαρτησία στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συμβάλλω για να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε τα μέλη του ε, Κοινοβουλίου να ασκήσουν αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο. Ε, ως γυναίκα θεωρώ ότι το, η διαφάνεια, η συμμετοχική ηγεσία, το να μοιραζόμαστε ε, απόψεις, το που γραζόμαστε τις απόψεις είναι αξίες πολύ σημαντικές και τις ενστερνίζομαι και θα ήθελα ε, αυτές τις αξίες να τις εφαρμόσω σε όλες τις επαγγελματικές και θεσμικές σχέσεις που θα έχω με εσάς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα πέντε τελευταία χρόνια ο χώρος δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισε πολύ σημαντική πρόοδο. Έχουμε τη δικαιοσύνη για τους πολίτες, τη δικαιοσύνη για την ανάπτυξη. Είναι πολιτικές αυτές που συνεισφέρουν με πολύ σημαντικές βελτιώσεις ε, την ε, καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, έχουμε την πρόταση για τις κληρονομιές. Θα διευκολύνει τη ζωή των οικογενειακών σε περίπτωση κληρονομιάς διασυνοριακής. Ε, με τον ίδιο τρόπο ένας Ευρωπαίος πολίτης εφ' εξής έχει τα ίδια δικονομικά δικαιώματα παντού στην Ευρώπη. Είτε πρόκειται για το δικαίωμα στη διερμηνία, είτε πρόκειται για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Από εκεί και πέρα έχουμε και προόδου σε θέματα πολιτική αστικού, αστικού δικαίου και εμπορικού δικαίου. Αυτά έχουν διευκολύνει τη ζωή των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το εξεκβάτουρ για παράδειγμα είναι κάτι το πολύ εύγλωτο, μιλάει από μόνο του. Καταργήσατε αυτή την επίπονη ε, δαπανηρή και μακροχρόνια διαδικασία αναγνώρισης δικαστικών υποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδείξει την ηγετική του θέση στα θέματα δικαιοσύνης, στα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, Εγώ έχω σημειώσει την εξαιρετική συνεργασία για όλα όλα αυτά τα θέματα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του τελευταίου Ιουνίου αναγνωρίζουν ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικές προόδους στην εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι η συνεργασία σε θέματα αστικά και ποινικά, αστικού και ποινικού δικαίου, ε, ευρωπαϊκή πολιτική σαν τις άλλες και έχουμε συναπόφαση. Αυτό είναι ο κανόνα. Άλλη μεγάλη προόδος και βελτίωση είναι η χάρτα των θεμελιδών δικαιωμάτων. Ε, αυτό το οποίο διακυβεύεται σήμερα είναι οι αξίες μας τις οποίες πρέπει να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε. Ε, η Ιταλική Προεδρία εξέφρασε σαφείς και φιλόδοξες ε, θέσεις για τους φακέλους μας και θέλει να προχωρήσουν οι φάκελοι σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εσείς είστε φιλόδοξοι και έχετε αναφερθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για θέματα προστασίας των δεδομένων. Είναι προτεραιότητα για τους επόμενους ε, μήνες. κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι να προετοιμάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τρίλογο, τον τριμερή διάλογο. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν εξαιρετική για το θέμα Τη προστασία των δεδομένων και χρειαζόμαστε τη στήριξή σας στους επόμενους μήνες. Έρχομαι τώρα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επεξεργασία των δεδομένων. Είναι σε καθοριστικό στάδιο. Έχουμε τη συμφωνία πλαίσιο, το Umbrella Agreement, ε, σε θέματα δικαστικής συνεργασίας και αστυνομικής συνεργασίας ε, και σε θέματα ανταλλαγής εμπορικών δεδομένων. Επομένως, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα ω προ την αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων δικαστική προσφυγή. για για τους Ευρωπαίους πολίτες κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης του περασμένου Ιουνίου και έχουν την πρόθεση οι ΗΠΑ να νομοθετήσουν για τα θέματα αυτά. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατυπώθηκε στην εξαιρετική έκθεση του κυρίου Μωράες και δεσμεύομαι να σας ε, ε, τηρώ ενήμερους για τις εξελίξεις ε, σε αυτό το φάκελο, οι οποίες με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Τώρα, έχουμε και το Safe Harbor, τον ασφαλή λιμένα είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την ανταλλαγή των εμπορικών δεδομένων. Έχει σημειωθεί πρόοδος και εκεί και είναι απαραίτητο ε, και οι 13 συστάσεις μας να υλοποιηθούν. Αυτές οι δύο διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο και για τον ασφαλή λιμένα είναι καθοριστικές για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με τις, Ηνωμένε Πολιτείες σε θέματα προσωπικών δεδομένων. Ε, έρχομαι τώρα στο θέμα της αφαιρεγγιότητας των επιχειρήσεων. Είναι, ένα, είναι κάτι που οι, οι προτάσεις μας για το θέμα αυτό είναι, κάτι που θα στηρί, είναι προτάσεις που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία. Ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα περιλαμβάνονται πλέον απαραίτητα στοιχεία για τη διάσωση των επιχειρήσεων και διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Και ελπίζω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έρθουν σε συμφωνία σε αυτό το στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ε, είναι ένα τεράστιο έργο με πολύ μεγάλη σημασία για το ε, μέλλον. Θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε την απάτη με πιο αποτελεσματικό τρόπο, να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι προτεραιότητα ε, για την ε, Ιταλική Προεδρία. Όπως επίσης και η οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης. Το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο έχει ήδη σημειώσει πρόοδο για τα δικονομικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη διερμηνία, το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα σε δικηγόρο και βασίζομαι σε εσά για να καθοριστούν και να θεσπιστούν ελάχιστα κοινά πρότυπα σε θέματα ποινικού δικαίου ω προ το τεκμήριο τη αθωότητα, την διαδικαστική και δικαστική βοήθεια, τι ε, δικονομικέ εγγυήσει υπέρ των παιδιών. Είμαι γυναίκα και είναι λογικό να προσδίδω ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος και για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και για οικονομικούς λόγους διότι έχει αποδειχθεί ότι ε, η εκπροσώπηση και των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και δεν είναι το μόνο, ε, ε το, ο μόνος ε, πάνω στον οποίο θα σημειώσουμε πρόοδο. Πρέπει να μην λησμονούμε σε καμία περίπτωση τον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας με την οποία υφίστονται οι γυναίκες, τον, ε, την καταπολέμηση των διακρίσεων που σχετίζονται με τα πιστεύω του καθενός και ε, την καταπολέμηση της υποκίνησης σε φιλετικό ή άλλο μίσος. Χρειάζεται να ε, μεριμνήσουμε ιδιαίτερως για τη δράση για την ένταξη των πληθυσμών Ρωμά και για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ε, ομοφιλοφίλων ανδρών, γυναικών φιλομεταβατικών ε, και λοιπόν. Ε, το να είμαι μέλος του Σώματος των Επιτρόπων θα μου επιτρέψει να συμβάλλω στην υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεσμεύομαι να προωθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ελεύθερη κυκλοφορία, ε, το κράτος δικαίου, την ισότητα όλων των πολιτών. Γνωρίζω τις προκλήσεις και θα αφιερώσω όση ενέργεια μπορώ για να τα φέρω σε πέρας με επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Very much, Ευχαριστούμε κυρία θα προβούμε τώρα στις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση από τον συντονιστή του ΕΛΚ για την Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών, κυρία Μόνικα Χολμά. 7 λεπτά συνολικά, παρακαλώ Μόνικα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κυρία Ράχερς, με την πρώτη ερώτηση. Καταρχήν μια ερώτηση που αφορά την προστασία δεδομένων. Συγκεκριμένα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται ότι αφενός ε, έχουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες που διαδραματίζουν ένα ρόλο κλειδιού για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε όμως το πρόβλημα ότι με το Google έχουμε ένα μονοπωλιακό, μια μονοπωλιακή επιχείρηση που όχι μόνο στρεβλώνει την αγορά και επιλέγει πληροφορίες τις οποίες ε, συλλέγει αλλά μεριμνά οι μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν ή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν στις αγορές χαρακτηριστικός ρόλος ενός μονοπωλίου, μιας μονοπωλιακής επιχείρησης. Ποιες προτάσεις ή ιδέες έχετε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Η Google για παράδειγμα να σέβεται το δίκαιο, ένα νομικό πλαίσιο ή να υπάρξει μια δικαιοσύνη όσον αφορά την λειτουργία των αγορών υπό αυτή την πτυχή. Σαν δεύτερο σημείο υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερες ανησυχίες έχουμε ότι οι μονοπωλικές επιχειρήσεις όπως η Google αντιμετωπίζουν τα δεδομένα ασίδωτα και επιβάλλουν τα κριτήριά τους στους καταναλωτές. Και γι' αυτό τον λόγο έχω την ερώτηση. Ποιες δυνατότητες βλέπετε να υφίστανται τέτοιου είδους μονοπωλικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα ασίδωτα και ελεύθερα όπως σκοπεύουν να το κάνουν και να υπάρχει μια δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και να συμμορφώνονται με το δίκαιο. Ένα άλλο θέμα για την αμοιβαία συνεργασία, αμφίδρομη συνεργασία, διασυνοριακά. Έχουμε διασυνοριακό έγκλημα ξεπερνά τα σύνορα αυτή η μορφή του εγκλήματος. Ερώτησή μου, πώς μπορούμε joint investigation teams, δηλαδή κοινέ ανακριτικές ή διακριβωτικές ομάδες να μπορούν με λιγότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση να συνεργάζονται και να δρουν άμεσα. Θα μπορούσατε να φανταστείτε μόνιμες ε, μορφές συνεργασίας ε, σε τέτοιου είδους ε, ομάδες που θα μπορούν μόνιμα να συνεργάζονται και να παρεμβαίνουν. Δεύτερον, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα για την αμοιβαία αναγνώριση των ανακριτικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά διασυνοριακές έρευνες ποιες μορφές, ας το αποκαλέσω έτσι, διεύρυνσης ή συμπλήρωσης υπό το ποινικό δίκαιο μπορείτε να φανταστείτε για την δίωξη σοβαρών εγκληματικών πράξεων διασυνοριακά. Τι θα προτείνατε. Μία ερώτηση και για την Όλαφα, την μονάδα καταπολέμησης απατών. Έχει αποδειχθεί ότι υπήρξαν παραβιάσεις και παραβάσεις και στις εξεταστικές δράσεις αποδείχθηκε ότι η Όλαφ σε σχέση με τον Γενικό Διευθυντή Κέσλερ για παράδειγμα και κάποιου άλλου αξιωματούχους σημειώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ρύθμισης ε, του κανονισμού 45-2001 και σε σχέση με την παραβίαση της ε, ιδιωτικής σφαίρας και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Θα είσαστε η αρμόδια επίτροπος στο μέλλον. Πώς θα καταφέρετε η Όλαφ και ο Γενικός Διευθυντής, η Διοικητής της Όλαφ και όλοι οι υπάλληλοι να σέβονται απόλυτα τα δικαιώματα του ανθρώπου και ε, να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πώς θα μεριμνήσετε και θα διασφαλίσετε ότι και η Όλαφ να συμμορφώνεται σε σχέση με αυτούς κανονισμούς. Μια τελευταία ερώτηση για την Eurojust σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μια και η Eurojust δεν πρόκειται να πάρει πρόσθετα κονδύλια αλλά άλλο έργο θα υποστεί ε, αρνητικές επιπτώσεις. Πώς θα διασφαλίσετε η εισαγγελία όχι μόνο να βρίσκεται στα χαρτιά αλλά να μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά της δημιουργώντας ένα πλαίσιο που με σάρκα και οστά θα μπορέσει να δράσει αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Και έτσι λοιπόν αυτές είναι οι ερωτήσεις από πλευρά του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω και θα επικεντρωθώ στην προστασία των δεδομένων. Στις 12 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο νομοθεσία στην πρώτη ανάγνωση και το διαβίβασε στο Κοινοβούλιο έκτοτε ε, στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη η Πολυνική Προεδρία ε, κατέληξαν οι Υπουργοί σε ένα προσωρινό πακέτο για την προστασία των ε, ατομικών δεδομένων και επίση συμφώνησαν για, το, για τη μόνο απευθυντική το τον ενιαίο τόπο εξυπηρέτησης. Ε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος ε, σε σχέση με το αρχικό κείμενο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο ε, από πλευράς περιεχομένου πώς θα, ακριβώς θα απομακρυνθεί από την αρχή της πρότασης Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε με ρεαλιστικό τρόπο και ευελπιστούμε και σύντομα να μπορέσει να εγκριθεί το πακέτο. Σε ποιο βαθμό οι συζητήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα για την ανταλλαγή προς προσωπικών δεδομένων εντάσσεται, πώς ακριβώς οι συζητήσεις αυτές θα επηρεάσουν το περιεχόμενο ε, των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για αυτό το πακέτο. Τώρα, σε σχέση με το πρόγραμμα παρακολούθησης NSA, ε, τον ΗΠΑ, επίσης στις 12 Μαρτίου ενέκρινε ε, το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το πρόγραμμα και την επιρροή που έχει επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί των διατλαντικών σχέσεων στον τομέα της δικαιοσύνης και των πολιτικών πολιτικών ελευθεριών. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα ούτως ώστε να ανακληθούν αμέσως οι ρήτρε σε safe harbor και ε, οι ερωτήσεις του εμπορικού επιμελητηρίου των ΙΠΑ ε, και να οριστούν νέες διατάξεις για τη μεταφορά ε, προσωπικών δεδομένων βάσει των απαιτήσεων των συνδικάτων σε αυτόν τον τομέα από ευρωπαϊκής πλευράς. Ποιες είναι οι προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα ζήτημα. Στο ίδιο ψήφισμα το Κοινοβούλιο επίσης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα νομική πρόταση για ένα νέο ε, σύστημα routing, ε, κυρίως ε, για τα λεπτομερή αρχεία που θα είναι μια υποδομή του ίντερνετ και δεν θα υπερβαίνει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς, τι είδους πρόταση θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστώ που δεν υπερβήκατε το χρόνο σας. Ε, η κυρία ε, είπε τώρα για ε, 6 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ράχερ, ζητούμε μία επίτροπο για ένα σχετικό σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό σε τρία θεματικά πλέγματα θα περιοριστώ. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω με τον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Το Ευρωκοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία διακομματικά διακοινοβουλευτικά έλαβε μια τέτοια απόφαση. Τροχοπεδήθηκε όμως η υπόθεση από το Συμβούλιο και γι' αυτό μας εξοργίζει αυτό ιδιαίτερα επειδή καθημερινά μέσω του διαδικτύου μπορούμε να διαπιστώσουμε νέες εξελίξεις που σημειώνονται και δεν έχουμε ρυθμιστικό πλαίσιο για όλα αυτά. Και είναι εξελίξεις ε, που αφορούν ε, και κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες ε, που εμπλέκονται. Πώς μπορείτε να φανταστείτε ότι η τροχοπέδηση του Συμβουλίου θα μπορούσε επιτέλους να αρθεί, να ξεπεράσουμε με το πρόβλημα. Σε αυτό το πλαίσιο φυσικά είναι σημαντικό η συμφωνία πλαισίου με τις ΗΠΑ για την ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά την θέματα ποινική δίωξη να ρυθμιστεί. Για μας είναι σημαντικό και λέγαμε ότι αν υπάρξει ποτέ μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει μια ρητή αναφορά για ένα μέσο νομικής αρρωγής και υποστήριξης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες δυνατότητες θεωρείτε ότι υπάρχουν ώστε μια τέτοια συμφωνία να μην πέσει πίσω από τις απόψεις, κάτω, να μην πέσει κάτω από τον γνώμονα και τον πύχη που θέτει το Κοινοβούλιο. Και ένας τελευταίος τομέας φυσικά για τα, τα δεδομένα είναι ο ασφαλής λιμένας, safe harbor. Για πολλούς συναδέλφους ευρωβουλευτές είναι μια αντίφαση στους ίδιους τους όρους αυτό, διότι δεν είναι ασφαλή αυτά τα δεδομένα. Και κάποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να καταγγελθεί αυτή η συμφωνία και να μην υπάρξει τέτοιο πλαίσιο. Η επανεξέταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που έγινε, είχατε ευκαιρία να εξετάσετε να δείτε ποιε εναλλακτικέ βελτιώσει θα μπορούσαν να υπάρξουν για αυτή τη συμφωνία ή αν υπάρχουν δυνατότητε πραγματικά εφόσον δεν μπορεί να λειτουργήσει να αποσυρθεί το, η πρόταση του ασφαλούς λιμένα και να υπάρξει μια άλλη ασφαλή διαδικασία. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της νομιμότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φυσικά στην υλοποίηση αυτό αποτελεί έργο των κρατών μελών. Οι αξίες μας όπως αντανακλώνται στις συνθήκες πρέπει να είναι σεβαστές όπως και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Να διασφαλίσουμε ότι στα κράτη-μέλη θα αποκτήσουν σάρκα και οστά αυτές οι ιδέες, αυτά τα ιδανικά. Έχει εδώ ένα πίνακα επιδόσεων, scoreboard η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει θεσμοθετηθεί, που έχει θεσπιστεί. Ωστόσο όμως και με το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Εξάμεινο ιδιαίτερα στον τομέα των ποινικών θεμάτων βρίσκονται στο περιθώριο. Εδώ στον τομέα του ποινικού δικαίου πρέπει σίγουρα να διασφαλίσουμε από πλευράς δικονομικών διαδικασιών ο σεβασμός της νομιμότητας και του δικαίου να διασφαλίζεται όχι μόνο όσον αφορά θύματα αλλά και οι υπόπτους ε, ή κατηγορουμένους. Ε, αναφερθήκατε στα δικονομικά δικαιώματα, στα διαδικαστικά θέματα. Ποιες δυνατότητες βλέπετε να μπορέσει να ασκηθεί πίεση ώστε αυτές οι αξίες για τις οποίες ε, εθελοντικά έχουν δεσμευθεί τα κράτη-μέλη σε όλους τους τομείς να μπορέσουν να επιβληθούν και να είναι σεβαστές αυτές οι αξίες. Και όχι μόνο στα χαρτιά να έχουμε αξίες και ζητήματα τα οποία διασφαλίζονται για τους πολίτες αλλά να είναι πραγματικότητα αυτά τα δικαιώματα. Και για τα θεμελιώδη δικαιώματα φυσικά άμεσα καταλήγουμε στο θέμα της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Σε πολλούς τομείς πολυσχηδός είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών, μεταναστών εργαζομένων, μειονοτήτων. Έχουμε μια στρατηγική για τους Αθηγάνους, τους Ρωμά. Πρόκειται όμως επίσης και για την αρνητική μεταχείριση και διάκριση με βάση τη θρησκεία και πολλά άλλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κάποιες οδηγίες επί των οποίων λόγους για αυτή την αρνητική μεταχείριση τους αναφέρουμε και απαγορεύουμε να υφίσταται τέτοια αρνητική μεταχείριση και διάκριση. Όμως βλέπουμε ότι σε συγκεκριμένους τομείς ε, όπως για παράδειγμα στην αγορά εργασίας ε, πρέπει κάτι να γίνει. Ε, απουσιάζει μια κοινή προσέγγιση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε αυτούς τους τομείς που θα απαγορεύει τις διακρίσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Έχουμε την εντύπωση ότι ένα τέτοιο ευρύτερο πλαίσιο ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση των ε, διακρίσεων αποτυγχάνει και τροχοπεδείται από πλευρά του Συμβουλίου. Έχουμε εδώ και το θέμα της τετραμηνίας που, που ε, έχει παρέλθει. Είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου ουσιαστικά. Μίζον πρόβλημα. Αλλά κάποιες ιδέες ε, έχετε για το τι μπορεί να γίνει ώστε να καταστεί σαφέστερο και να πιεστεί το Συμβούλιο να αναλάβει περαιτέρω δράση και να προαγάγει αυτά τα θέματα ώστε να προοδεύσουν. Αυτά είναι θέματα από τις ερωτήσεις που θέλαμε να σας διατυπώσουμε. Ευχαριστούμε, Μπριγκίτ. Εντάξει, είναι για λίγους μήνες. Φύγετε από τώρα, άμα θέλετε. Όχι, αστείευομαι. Μπορείτε να κάτσετε φυσικά από τον συντονιστή του ECR, Τίμωθη Κυρκόπ. Καλώς ορίσατε κύριε Ρέχατ στην ακρόαση μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στις παρατηρήσεις κυρίας Χόλμαγκερ για τις GIS, τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες, διότι ήμουν εισηγητής για αυτή την πρόταση εδώ στο Κοινοβούλιο και με απογοητεύει το ότι δεν έχουμε φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας σε επίπεδο ερευνητικών ομάδων στην Ευρώπη. Ε, τώρα, ε, ε, λόγω της ανησυχητικής και σταθούς κατάσταση στη Συρία και στην, στο Ιράκ και λόγω της δράσης Ισλαμιστικών ομάδων όπως η ΙΣΙΣ ε, μπορείτε να μας πείτε ε, στα πλαίσια της αστυνομικής συνεργασίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ένα θέμα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Μπορείτε να μας πείτε αν πιστεύετε πως η μεταρρύθμιση και ε, το άνοιγμα εκ νέου του πακέτου αυτού είναι προτεραιότητα στον τομέα της δικαιοσύνης και των ε, πολιτικών ελευθεριών. Θα ήθελα να αναλυφθεί η από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνα. Ε, μπορεί να είναι χρήσιμο το εργαλείο, αλλά χρειάζεται ε, ε, να, οπωσδήποτε να μεταρρυθμιστεί άρδιν. τώρα, Το δικαίωμα λίδης τώρα για την, ε, ε, ε, την διαγραφή των δεδομένων σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μάθαμε ότι διάφοροι πολιτικοί ζήτησαν εκ των υστέρων να διαγραφούν άρθρα για προηγούμενες αξιόπινες πράξεις. Επαγγελματίες ζητούν να διαγραφούν από τα αρχεία παλαιότερες υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ασαφές είναι και δεν οδηγεί οδηγεί σε καταλητικά συμπεράσματα χωρίς τη δέωσα νομοθεσία. Αν δεν ξέρουμε τι είναι και τι δεν είναι προς, συμφέρον, ε, προς ε, το κοινό συμφέρον, πώς μπορούμε να παίρνουμε οποιασδήποτε αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Ε, ε, Τιμωθή, μπορείτε να απόσχετε από την απάντηση σε ερωτήσεις όπως αυτή για τη γιόγκα. Τώρα θα ακούσουμε για δύο λεπτά τη Σεσίλια Μάλμστρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την υποψήφια Επίτροπο. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ένωση αν δεν υπάρχει ένα σύνολο Ευρωπαίων πολιτών με κοινέ αξίε και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι η πλατφόρμα για τη συνεργασία και για μια εύρυθμα λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, θα, δείξετε, θα επιδείξετε την απαιτούμενη αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των διατάξεων προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αν χρειαστεί ακόμη και να αναλάβετε δράση κατά των κρατών μελών που δεν σέβονται τις ε, νομικές διατάξεις σε σχέση με το κράτος δικαίου και τα θεμελιωδία δικαιώματα. Ε, τώρα για τις διαδικασίες σε παραβάση για τα, εναντίον των κρατών μελών για παραβίαση ε, του κράτους δικαίου και θεμελιωδών ελευθεριών όπως παραδείγματος χάρη πολιτικές ελευθερίες, ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, δικαιώματα των Ρωμά, δικαιώματα των ΛΟΑΔ και ούτω καθεξή Θα αναλάβει τέτοια δράση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν θα ενισχύσετε το καλό έργο της κυρίας Τρέντινγκ για την ε, μεταρρύθμιση του πίνακα επιδόσεων του ώστε να καλύπτεται το κράτος δικαίου και ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και ευρύτερα και ένα πιο προσωπικό σχόλιο. Ποια πρόταση θα κάνετε για περαιτέρω παρακολούθηση ε, της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σισίλια. Από πλευράς του ομάδας EFTD, κυρία Λάουρα Φεράρα, για ένα λεπτό. Καλησπέρα σας, κυρία Ράιχερτς. Ξέρετε, μια χώρα τη θεωρούμε πολιτισμένη από τη στιγμή που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της και αναφερόμαστε σε δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε ανθρώπινο όν που διαβεί μέσα στη δική μας κοινωνία. Ωστόσο, ε, πολλοί ε, στερούνται αυτών των δικαιωμάτων και εκεί έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και αναφέρομαι σε κάποια ελάχιστα πρότυπα συνθήκων κράτησης και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ κρατών μελών για το θέμα αυτό. Γνωρίζετε ότι ε, κάποια κρατημέλη πόρο απέχουν από το να είναι σε θέση να εγγυώνται ανθρώπινες συνθήκες κράτησης για τους ανθρώπους αυτούς και υπάρχουν συνθήκες κράτησης οι οποίες ισοδυναμούν με βασανιστήριο. Πρόκειται για απάνθρωπη και εξαθλιωτική μεταχείριση ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπλακεί στα δίχτυα αυτού του συστήματος της τιμωρίας. Ε, είναι άνθρωποι που στρέφονται προς την αυτοκτονία και γι' αυτό έχουμε τόσο σημαντικά ποσοστά αυτοκτονιών άλλωστε είναι άνθρωποι που υποφέρουν ε, και χρήζουν άμεσης ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα για τους κρατούμενους και θα πρέπει να αναδιατυπώσουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενες ερωτήσεις από πλευράς Γκουε. Η κυρία Κορνίλια Έρτστ, για ένα λεπτό. Γεια. Μάλιστα. Και από εμά καλωσορίσατε θερμά κυρία Ράχες. Χαιρόμαστε ότι έχουμε αυτή τη διαδικασία που ξεκινά. Έχουμε ρωτήσει όπως για τα δεδομένα, προσωπικά δεδομένα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής, ποιο είναι το δικό σας χρονοδιάγραμμα. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι επίσης και το Συμβούλιο, πώς να το πω, την τροχοπέδηση αυτή σε σχέση με την οδηγία, όχι μόνο τον κανονισμό αλλά και την οδηγία θα την αντιμετωπίσουμε. Επίσης το δεύτερο θέμα είναι η κατασκοπία εις βάρος πολιτών της Ευρωπαϊκής, ε, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια διαβήματα θα κάνετε για τις παραβιάσεις της NSA, της ε, Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ με κατασκοπία πολιτών. Είναι θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που παραβιάζονται. Τρίτο σημείο, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζονται. Το βλέπουμε αυτό και σε άλλες χώρες. Έχουμε και μια έκθεση για την Ουγγαρία, την έκθεση Ταβάρες, έχουμε και την έκθεση Μισελ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ερώτησή μου είναι, τι έχετε υπόψη σας να πράξετε στην υλοποίηση αυτών των μέτρων που πρέπει να προαχθούν. Και τελευταίο, μια εξαιρετική στρατηγική για τους Ρωμά, τους Αθηγάνους. Όμως ποτέ δεν ήταν τόσο έντονη η διάκριση, η διακρίση εις βάρος των Τσιγκάνων όπως ε, πρόσφατα. Τι θα κάνετε ώστε να υπάρξουν πιο δεσμευτικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούνται ώστε να αρθεί να αντιμετωπιστεί η διάκριση εις βάρος των Ρώμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από τους Πρασίνους, ε, ε, Σαρτζεντίνη. Α, ο Γιάνν Άλμπρεχτ θα την αντικαταστήσει κυρία Σατζέντινη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία, κυρία Ρέχερ, σε τρει ερωτήσει έχουμε από τον Απρίλη προς το, μέχρι τον Ιούνιο. 4.000 ε, Ρωμά ε, ε, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το, γαλλικό έδαφο. Ε, Πώ σκοπεύετε να προστατεύσετε τα θεμελιώδη δικαιώματά του. δεύτερον, ο Οργανισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και διακριτική μεταχείριση κατά τον ΛΟΑΤ και τον αντισημιτισμό ε, κάνει μελέτες που δείχνουν ε, ένα πάρα πολύ ε, κακό κλίμα σε σχέση και με τα εγκλήματα μίσους. Το 2008 έγινε μια πρόταση για αυτά τα εγκλήματα που πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά δεν δόθηκε συνέχεια. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να πιέσετε τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να εγκρίνουν αυτό το νομοθέτημα που, που προτείνετε. Στη συνέχεια τώρα δεν θα μπω εγώ στα προσωπικά δεδομένα γιατί ακούσαμε ήδη πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να τα πω μόνο ότι πέρα από την απόφαση για το Google υπήρξε και μια απόφαση για την ε, ε, παρακράτηση δεδομένων και ε, υπάρχει και η οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτική σφαίρα που εντάσσεται στο πακέτο της ασφάλειας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Υπάρχουν δράσεις που παρεβιάζουν αυτή την απόφαση, καθώς και διατάξεις οδηγίας για την ηλεκτρονική ιδιωτική ζωή, ε, θα κινήσετε διαδικασίες σε παραβάση κατά των κρατών μελών παραβιάζουν αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστούμε Γιάννη. Ε, ολοκληρώνεται έτσι ο πρώτος γύρος ερωτήσεων των συντονιστών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές διότι δεν επιρβήκα το χρόνο ε, αγόρευσης που σας αναλογεί και χάρη σε αυτό ε, λόγω της αρχής καθυστέρησης κερδίσαμε χρόνο. Ευχαριστώ για την ποιότητα των ερωτήσεών σας. Πραγματικά αυτά τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων είναι κέρια σημασία για την Επιτροπή Πολιτεχνικών Ελευθεριών. Κυρία Ράιχερτ, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού τα υπόλοιπα 10 10 λεπτά, τα επόμενα συγγνώμη 10 λεπτά να απαντήσετε ε, σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τι ήταν έργο μου ζητάτε να κάνω. Δεν μου φτάνουν τέσσερι μήνε που θα είναι η θητεία μου, αλλά τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Σε κάθε περίπτωση σα ευχαριστώ θερμά για όλε αυτέ τι ερωτήσει και θα προσπαθήσω να τι ομαδοποιήσω τρόπον Α και σα ζητώ συγγνώμη διότι δεν θα προλάβω να μπω σε λεπτομέρειε σε κάθε μία ναι. ερώτηση γιατί 10 λεπτά είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αλλά ελπίζουμε ότι θα βρισκόμαστε πιο συχνά και θα είμαστε σε θέση τότε στι επόμενε συνεδριάσει μα συνεδριάσεις μας και συναντήσει μα να βγούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Να ξεκινήσω από τα προσωπικά δεδομένα γιατί είναι και το πιο, ε, ο πιο σημαντικός φάκελος ο οποίο βρίσκεται επιτάπητο αυτή τη στιγμή. Βλέπετε πόσα προβλήματα ε, έχουν δημιουργηθεί με τι ΗΠΑ, την Google, τη Microsoft και ούτω καθεξής. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δομήσω την απάντησή μου έτσι ώστε να καλύψω διάφορες ερωτήσεις από τους ερωτώντες. Σας ευχαριστώ όλους θερμά γιατί δείχνετε πόσο σας ενδιαφέρει ο φάκελος αυτός. Είχαμε μια μερική συμφωνία στο Συμβούλιο της 6ης Ιουνίου και τι προτίθεμαι να κάνω. Η κυρία Ζήπφερ νομίζω το ρώτησε αυτό. Μεγάλη πρόοδος επιτεύχθη στο άτυπο συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας, ενδεχομένως κάποιοι από εσά είσαστε παρόντες και έγινε συζήτηση για την ευελιξία για τον δημόσιο τομέα σε αυτόν τον κανονισμό. Και ήταν μια συζήτηση που προχώρησε ιδιαίτερος. Ξέρω ότι ήταν μεγάλο το πρόβλημα για τις γερμανικές αρχές και έτσι η μερική συμφωνία της περασμένης εβδομάδας στο άτυπο συμβούλιο διευκόλυνε την κατάσταση και θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ε, μέχρι το τέλος της χρονιάς ίσως το προλάβω και εγώ. Αναφέρα, αναφερθήκατε στην Google, αλλά υπάρχει και η Microsoft και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς και επιθετικούς προσδιορισμούς για αυτές τις δύο εταιρείε. Σε κάθε περίπτωση έχουμε απέναντί μας εταιρείε που έχουν αντιφατικές υποχρεώσεις. Ε, το νομικό καθεστώς στις ΗΠΑ δεν είναι το ίδιο με το δικό μας. Έχουμε σεβασμό δικαιωμάτων στην Ευρώπη από τη μία και από την άλλη οι Αμερικάνοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν εξετάσει αυτό το θέμα επανειλημμένος και δεν θα σας εκπλήξει ε, ε, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένως έχει πει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να διαβιβάζονται ή να είναι άμεσα προσβάσιμα παρά μόνο στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών οι οποίες υφίστανται αυτή τη στιγμή και ε, πιο συγκεκριμένα η συμφωνία πλαίσιο Umbrella Agreement. Να επανέλθω στο νομοθετικό πλαίσιο έτσι όπως προτάθηκε και να πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της του 2012 έχει ενισχύσει το εξής σκέλος. Οι εταιρείε που λειτουργούν στην Ευρώπη οφείλουν να σέβονται ε, τα, ε, τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε θέματα προστασίας δεδομένων. Και άρα εδώ έρχομαι σε στην απάντηση στην κυρία Μάγερ και θα πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατό όλη αυτή τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων. Δύο λόγια να πω ε, για την Google. Και εγώ όπως και εσείς διάβασα τις εφημερίδες το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ σημαντικός ο φάκελος αυτός. Δεν μπορώ να ε, το σχολιάσω το θέμα ξεκάθαρα σήμερα γιατί συνεχίζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύουμε διάφορα δεδομένα η λέξη κλειδί είναι η λέξη ισορροπία ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση και των δικαιωμάτων των ατόμων για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνάδει με την απόφαση του δικαστηρίου και ε, σε σχέση με τον Γιάνν Άλμπρεχτ και ε, ε, παρακαλώ να μας δώσετε λίγο χρόνο ως προς τη διαφορετική στάση των κρατών μελών έναντι της νομολογίας του δικαστηρίου και θα πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη υπό το φως ε, της απόφασης του δικαστηρίου. Ε, για μένα λοιπόν η λέξη κλειδί είναι η λέξη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο πολύ σημαντικών στοιχείων. Ως προς τον ασφαλή λιμένα, το safe harbor και με, για αυτό το θέμα μίλησα με τον κύριο Άλμπρεχτ, σημείωσα ότι ζητείτε την αναστολή όλων αυτών, το μήνυμά σας είναι σαφές. Ωστόσο, η Επιτροπή το Νοέμβριο του 2013 είχε δημοσιεύσει 13 συστάσεις και έκτοτε ε, είναι σε διαπραγμάτευση η κυρία Λεμπάγ ε, είναι στην αίθουσα εδώ, είναι στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Γίνονται λοιπόν συζητήσεις, εκτιλήσονται οι συζητήσεις και η κυρία Λεμπάγ, δεν τους έχω συναντήσει ακόμα, δεν είχα χρόνο. Ε, με διαβεβαίωσε όμως η κυρία Λεμπάγιο ότι η πρόοδος είναι σημαντική, ειδικότερα ως προς τα θέματα διαφάνειας. Και σας υπενθυμίζω ότι ξεκάθαρη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το φάκελο είναι η εξής. Ζητούμε από τους Αμερικανούς να ελοποιήσουν και τις 13 συστάσεις. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν και νομίζω ότι η Φρανσουάς Λεμπάγιο θα έρθει να σας τα εξηγήσει αυτά. Ε, αν δεν είναι αυτή τη βδομάδα θα είναι την επόμενη εβδομάδα να σας εξηγήσει την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και όταν θα ε, σας συντάξει μια ξεκάθαρη έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τη διαπραγματεύση αυτό το φάκελο μπορείτε να μας υποβάλλετε τις απόψεις σας γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Τώρα, ως προς τις ανάγκες για θέματα εθνικής ασφαλείας μιλούμε για μια αρχή εξαίρεση με την επίκληση των λόγων της εθνικής ασφαλείας στο πλαίσιο του ασφαλή λιμένα του Safe Harder είναι μια εξαίρεση η οποία θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό. Μόνο εξαίρεση. Πρόκειται για αρχή δικαίου. Τώρα, το, οι συμφωνίες Umbrella. Να πω δύο λόγια. Και εδώ έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Αμερικανικών αρχών, οι οποίες δεσμεύτηκαν να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων όπως και οι Αμερικανοί πολίτες. Και αυτό πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και οι διαπραγματεύσεις που εκτελήσονται πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Επομένως, έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, αυτά με τα προσωπικά δεδομένα, στην ελεύθερη κυκλοφορία. Και εσείς το επαναλάβατε και εγώ θα το επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω μάλλον όσο μπορώ, η ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Είναι μία από τις τέσσερις τεράστιες θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πυλώνας δικαίου και πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλα αυτά. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ωστόσο, ε, διάφορα κινήματα υπάρχουν ε, και κινήσεις υπάρχουν στα κρατη ε, και θα πρέπει πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πρέπει η προσέγγιση μας να είναι ρεαλιστική με σκοπό τον περιορισμό των καταχρήσεων. Π.χ. το εχειρίδιο για τους γάμους συμφέροντος, ε, τους λευκούς γάμους, γιατί πρέπει να το πούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και έχουμε εχειρίδιο για αυτό. Τώρα, ως προς το φάκελο για τα δικαιώματα λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αμφιφιλοφίλων, φιλομεταβατικών. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διακρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Έχουμε οδηγία για την, ε, την αρχή περί μη διάκρισης και βεβαίως εφαρμοστέως είναι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και δεσμεύω προσωπικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτός ο φάκελο. η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, που έχει εγκριθεί, να εφαρμόζονται πλήρως και επί της αρχής και επί της ουσίας έτσι ώστε και αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες να ε, μπουν σε αυτή την κατηγορία. Ε, δεν είναι το θέμα ε, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μιλούμε μόνο για την απομόνωσή τους. Είναι πολύ περισσότερο και πολύ σημαντικότερο από αυτό. Δεσμεύομαι λοιπόν να κάνω το παν έτσι ώστε να εγκριθεί η οδηγία που έχει να κάνει με το άρθρο 19 και για τη μία μη διάκριση, αλλά δεν χρειάζεται σε εσά, Γιάνν Άλμπρεχτ, να πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Το γνωρίζετε και γι' αυτό βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη. Τώρα, ως προς τους ε, πληθυσμού Ρωμά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί προσπαθεί να υιοθετήσει θετικά μέτρα. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα στα κράτη-μέλη και πρέπει να ακούσουμε τα κρατη και τους πολίτες. Ωστόσο η ελεύθερη κυκλοφορία παραμένει αρχή και είναι σημαντικό να φτάσουμε σε ένα σωστό σημείο ισορροπίας και εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσέγγιση της επιμένει για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά να έχουν πρόσβαση στις, στο σχολείο, στις υπηρεσίες υγείας, στην απασχόληση. Αυτό είναι θεμελιώδες γιατί εάν ενταχθούν κοινωνικά και όποτε εντάσσονται κοινωνικά πάρα πολλά προβλήματα ρυθμίζονται και επιλύονται. Ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θέματα ποινικού δικαίου. Εξαιρετικά σημαντικός αυτός ο φάκελος επίσης, όπως μας το υπενθυμίσατε, θα έχουμε όργανα ε, τα οποία θα λειτουργούν σε σώμα ε, με εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη και θα συνεργάζονται με τα υφιστάμενα θεσμικά ε, όργανα. Δηλαδή δεν αφαιρούμε τίποτα, δεν κατερκούμε κανέναν φορέο, φορέα και τονίζουμε την ιδιαιτερότητα του ποινικού δικαίου στο κάθε κράτος μέλος. Τι έχω ξεχάσει. Ο υπερπληθυσμός στις ε, φυλακές, η συσσόρευση στα σοφρονιστικά ιδρύματα, η κυρία Φεράρα έθεσε το σχετικό ερώτημα και πράγματι είναι σημαντικός ο φάκελος αυτός και είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή είναι ασύμβατη με το τεκμήριο της αθωότητας, μια αρχή, γενική αρχή δικαίου για τους νομικούς και θα προσπαθήσουμε όσο θα το πιο γρήγορα να υλοποιήσουμε τις τρεις αποφάσεις πλαίσιο για τις συνθήκες κράτησης τις οποίες ασωματώνουν αυτή τη στιγμή τα κρατη στην εσωτερική τους νομοθεσία για να περιορίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Αυτά κύριε Πρόεδρε, δεν έχω άλλο χρόνο από ό,τι βλέπω. Είμαι έτοιμη να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις ή να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες είτε στη συνέχεια είτε μετά τη λήξη της ε, συνεδρίασης ε, ατομικά ε, με τον καθένα από εσά, αλλά αν ανάψει και δεύτερο κόκκινο αστεράκι νομίζω ότι θα με ψέξει ο Πρόεδρος γιατί θα έχω καθυστερήσει πολύ. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ερχόμαστε τώρα στις ερωτήσεις από πλευρά συντονιστών της Επιτροπής Γιούρη κύριου Σιβκέφκα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θαυμάζω πραγματικά την ε, συντομία στην έκφρασή σας ε, και το ότι τηρήσατε το χρόνο όντας τόσο σύντομη. Πέρα από αυτό θα ήθελα δύο παρατηρήσεις να διατυπώσω. Η Σεσίλια Βίστρομ ήδη ανέφερε ότι η οικοδόμηση μιας ισχυρής ένωσης πρέπει να βασίζεται σε κάποιες κοινέ αρχές και αξίες. Θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτό ότι πρέπει να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια παράδοση νομική κοινή για την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά κράτη και αυτό συζητούμε επί αρκετό διάστημα στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή ως θέμα. Τώρα σε σχέση με τις αποφάσεις την ομολογία του δικαστηρίου όσον αφορά εμπορικά θέματα και την υιοθέτηση λύσεων. Και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει να τηρούνται και να είναι σεβαστές στα κράτη-μέλη. Τον ε, Ιούνιο <clears throat> το Συμβούλιο ζήτησε να ενισχυθεί η αποφασιστικότητα και το σθένος μας ε, προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει ανάγκη αναλλαγή ε, στοιχείων και πληροφοριών για τα νομικά μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα πλέον τώρα και είναι στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρηματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η ερώτησή μου, ποια βήματα και διαβήματα θα κάνετε ώστε να ενισχυθεί αυτό το μέσο, να ενδυναμωθεί και να μπορέσουν αυτά τα μέτρα να καταστούν πιο προσπελάσιμα και καλύτερα, ε, πιο εύκολα στη διάθεση των ε, επιχειρηματιών. Και για την νομική, το νομικό, την νομική παράδοση και πλαίσιο που πρέπει να υιοθετηθεί και να λειτουργήσει χρειάζεται εμπιστοσύνη, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και για να γίνει αυτό πρέπει να μπορέσουμε να καταρτήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους δικαστές και τους εισαγγελείς ε, από πλευράς δηλαδή της δικαστικής εξουσίας με τον κατάλληλο τρόπο. Πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα πρόγραμμα πιλωτικό ε, ε, θα θέλαμε να μας εκφράσετε τις δικές σας απόψεις ε, υπό αυτό το πρίσμα. Κατά ποιο τρόπο αυτά τα μέσα θα μπορούσαν να ενδυναμωθούν, να ενισχυθούν περαιτέρω και να λειτουργήσουν καλύτερα. Και μια άλλη παρατηρήση αν επιτρέπετε αφορά το νόμο, το πλαίσιο για τις πωλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια χρόνια πριν, τρία χρόνια πριν, το 2011 τον Ιούλιο, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού νομικού πλαισίου όσον αφορά το δίκαιο για τις πωλήσει ε, ε, Πρέπει να πούμε ότι ε, έχει προχωρήσει το έργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ δυστυχώς στο Συμβούλιο αυτό λιμνάζει. Η εικόνα είναι απεσιόδοξη έτσι όπως αντανακλάται από το Συμβούλιο. Ε, από πλευρά εισηγητού που δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας θα πρέπει να διορίσουμε νέους εισηγητές. Ερώτησή μου, θα υποστηρίξετε τις δράσεις αυτών των εισηγητών προς αυτή την κατεύθυνση, τις δραστηριότητες τους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να στεφθούν επιτυχία αυτά τα εγχειρήματα. Είσαστε υπέρ αυτής τη εναλλακτικής λύσης, εναλλακτικού δηλαδή πλαισίου για το δίκαιο πολίσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ρέγνερ, τώρα 3,5 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ η κυρία Ρέγνερ. Καλωσορίζουμε την κυρία Ράιχερτς και για το γεγονός ότι πιέζει ο χρόνος θα επικεντρωθώ αποκλειστικά σε εκείνα τα θέματα που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά για μας και έτσι θα επικεντρωθώ σε κάποια ξεχωριστά θέματα που έχουμε υπό εξέλιξη. και οι ερωτήσεις μου θα επικεντρώνονται σε αυτά τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι σημαντικό για τους πολίτες μας να βρισκόμαστε πολύ κοντά στις ανησυχίες και τα μελήματα των πολιτών, να απλουστεύσουμε τα πλαίσια των νομικών εγγράφων που χρειάζονται από πλευρά των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω υποψήφια επίτροπο, θα γνωρίζετε ότι σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωκοινοβούλιο καλωσόρισε αυτή την προσέγγιση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απλούστευση και την αποδοχή των νομικών εγγράφων. Καθώ επίση και την εξειδίκευσή του ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά. Η Επίτροπο Ρέντινγκ επικεντρώθηκε σε αυτά τα θέματα με ιδιαίτερο σθένος. Ερώτησή μου, ποια είναι η άποψή σας σε σχέση δηλαδή με τις ε, ε, πιστοποιημένες μεταφράσεις ε, και τέτοιου είδους απαιτούμενα έγγραφα. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα εξειδικευμένα και κυρίως επίσης για την αναγνώριση όσον αφορά τα έγγραφα που αφορούν τους πολίτες και το καθεστώς τους Επίσης ε, η δεύτερη παρέμβασή μου αφορά την παρέμβαση του κυρίου Σβιεύκα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα διέπει τις πωλήσει ε, νομικά. Ερώτηση, τι μπορείτε εσείς να κάνετε ως υποψήφια επίτροπος, ε, τι θα κάνετε πραγματικά ως αρμόδια για αυτό το χαρτοφυλάκιο πιο εξειδικευμένα. Το τρίτο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και επιλέγω, το αναφέρατε στην εισαγωγή σας ήδη το θέμα για την αντιμετώπιση πτωχεύσεων στην πρώτη ανάγνωση απέτησε το Κοινοβούλιο ότι περαιτέρω μέτρα πληροφόρησης και εναρμονισμού θα πρέπει να προβλέπουν προτιμησιακά δικαιώματα για αυτές τις περιπτώσεις. Υποστηρίζεται αυτή την ιδέα και θα αντανακλάται στις μελλοντικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έρχομαι και σε μια ναυαρχίδα ως θέμα της ε, Αντιπροέδρου ε, κυρίας Ρέντινγκ τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και θα πρέπει εδώ να δούμε και τι γίνεται με εταιρείε ε, που δρούν στα χρηματιστήρια παρότι υπήρχαν κάποιες διαφορές σε σχέση με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμείς αυτά που αποφασίσαμε και εγκρίναμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δεδομένα. Η κυριότερη διαφορά σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι <clears throat> η ε, διαγραφή ή μη δυνατότητα να συνεχίσουν ε, ε, να λειτουργούν αυτά τα συμβούλια όταν θα βρίσκονται οι γυναίκες και θα εκπροσωπούνται κάτω από το 10% των μελών. Θα δώσετε συνέχεια σε αυτή την ιδέα πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποστηρίξαμε στο μέλλον. Μία άλλη πτυχή που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το θέμα των κυρώσεων. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα πίνακα κυρώσεων που έχει αποφασίσει και εγκρίνει και την α, τον αποκλεισμό από την υποβολή ε, προτάσεων για δημόσιες προμήθειες ε, και ε, συμβάσεις. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού του θέματος και εν τέλει με ποιο τρόπο αντιμετωπίζετε εσείς σε σχέση με τα θέματα τα οποία εκκρεμούν με το Συμβούλιο και με εκείνες τις χώρες ε, που έχουν μια κάπως ε, πιο ουδέτερη θέση επ' αυτού. Τι θα πράξετε ώστε να διευρυνθεί, ας το πω έτσι, το πλαίσιο συνένεσης, ώστε να προαχθεί το θέμα και να οριμάσει και να ολοκληρωθεί από πλευρά διαδικασιών και ώστε αυτές οι διαδικασίες να στεφθούν με επιτυχία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρίμα από την ECR. 1,5 λεπτό. Σας καλωσορίζω κυρία Ρέχας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι σύντομη η θητεία σας, αλλά είναι κέρια σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή κατάσταση αυτή τη στιγμή που μας κοιτάζουν όλοι και περιμένουν ανάπτυξη. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτε της. Πώς βλέπετε ακριβώς τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, κυρίως ε, σε σχέση με την απάντηση της κυρίας Ρεντίνγκ ε, για τα θέματα Επικουρικότητα για το θέμα τη εισαγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνω υπόψη αυτά που μα είπατε στις αρχικέ δηλώσει. σα. Συμφωνείτε με την άποψη ε, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και της Ολομέλειας ότι δηλαδή ο διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβουλία θα πρέπει να αναβαθμιστεί και βάσει μελετών θα πρέπει να διερευνηθούν οι μέθοδοι ενίσχυση ε, του μηχανισμού επικουρικότητα και δεύτερον, και τώρα στρέφομαι προ ε, το θεματολόγιο το αναπτυξιακό, ε, επιχώντας ε, και τα ζητήματα που ήγηραν ε, οι δύο συντονιστέ ε, για το κοινό εταιρικό δίκαιο, δίκαιο πολίσεων, συγγνώμη, θα ήθελα να σας καλέσω να προβληματιστείτε για το εξή. Πέρα από τους εμπλεκόμενους φορείς, οι εθνικές κυβερνήσεις, εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γίνουν ερωτήματα σε σχέση με την σκοπιμότητα των προτάσεων. Η νομοθεσία, όπως παραδείγματος χάρη μικρές αξιώσεις δικαιώματα καταναλωτών και ε, συναφή νομοθετήματα που τώρα αρχίζουν να εφαρμόζονται και μπορούν ενδεχομένως να έχουν θετική επιρροή σε σχέση με την ε, διασυνοριακή δυνατότητα συναλλαγών για τους ε, ιδιώτες και για τις επιχειρήσεις. Μήπως θα έπρεπε καλύτερα να βελτιώσουμε την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σημειώνω ότι δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε επίσης νεότευκτα μέτρα και πώς, ε, ποιες είναι οι εξελίξεις που προβλέπετε και είναι κυρία σημασία για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς και δεν αναφερθήκατε σε αυτό, πώς είσαστε εσωστρεφείς αντί για εξωστρεφείς. Σας ευχαριστούμε. Κύριε καρίμο ο κύριος Καβαντά τώρα από πλευράς ε, των φιλελευθέρων 1,5 λεπτό. Θα ήθελα... Καλώς ήρθατε κυρία Ράιχερτ. Με δεδομένο το προφίλ σας, Πρέπει να σας πω ότι είμαι ο πιο κατάλληλα τοποθετημένος για να σας πω ότι έχετε πολύ σωστό αξίωμα. Είστε ο κατάλληλος άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Από εκεί και πέρα ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για την εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα ε, γάμων, για την κληρονομιά, για τα κληρονομικά δικαιώματα, για την επίπτωση που έχει η σύναψη γάμου ε, στην περιουσιακή κατάσταση των ατόμων. Περιμένουμε σχετική απόφαση του Συμβουλίου εδώ και καιρό. Η Επιτροπή στην οποία ανήκω στο παρελθόν έχει απευθύνει έκκληση για την αμοιβαία αναγνώριση των υιοθεσιών. Γιατί είχαμε περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Επικράτειο όπου οι γονείς που υιοθέτησαν άλλαξαν χώρα, μετήκησαν σε άλλη χώρα και τους απέσυραν, τους πήραν τα παιδιά τους γιατί δεν τους είχε αναγνωριστεί το καθεστώς του ε, γονέα που υιοθετεί παιδί. Επομένως, η αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης, των ε, συμφώνων συμβίωσης, όλα αυτά θα γίνουν επιτέλους. Ε, η αμοιβαιότητα δηλαδή όλων αυτών των αποφάσεων και ε, θα, έχουν, θα γίνουν και για το θέμα των υιοθεσιών όπως το έχουμε συζητήσει και ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να αναφερθώ τέλος και σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Είναι απαραίτητο τα κράτη που δεν εφαρμόζουν τον χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων να ε, υφίστανται κυρώσεις και όχι μόνο προειδοποιήσεις. Το οποίο έκανε η προκάτοχό σα δεν είχε τα πολιτικά μέσα να κάνει ε, να επιβάλλει κυρώσεις παρά μόνο προειδοποιήσεις αφιερώσετε την ενέργειά σας ε, αγαπητή κυρία για να, να ξαναγίνουν αυτά τα οποία είχαν γίνει με την Αυστρία και είδατε πόσο ωφέλησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγονος από την πλευρά της ΓΚΟΕ για 1,5 λεπτό. Okay. Not Δεν είναι παρόν. Η κυρία Χάουτα από τους Πράσινους για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ράχερτς, έχω δύο ερωτήματα να σας απευθύνω. Το πρώτο για τη διατησία, η οποία έχει γίνει θέμα και στην ευρύτερη δημόσια συζήτηση λόγω ε, της ε, ε, συμφωνίας ε, διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, εταιρικής σχέσης για όλα αυτά. Είχαμε λοιπόν τον κανονισμό Βρυξέλλες 1, τον αναθεωρημένο, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ ήδη εδώ και αρκετό καιρό και ε, υποτίθεται ότι θα αποκλειόταν η διαιτήση από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού. Ωστόσο αυτό έδωσε λαβή για ασάφειες. Ερωτώ λοιπόν το εξής. Συμφωνείτε ότι ε, για να δοθεί προτεραιότητα ε, στα, ε, στο δικαστικό σύστημα του κράτους σε περίπτωση διαιτησίας πρέπει να ε, ξεκαθαριστεί περισσότερο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται διαιτησία και που να ξεκαθαριστεί στο σχετικό κανονισμό Βρυξέλλες 1. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω για τις οικογένειες και για τα παιδιά. Πού ε, γνωρίζετε τη συζήτηση που γίνεται ε, στο Συμβούλιο. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τη Σύμβαση της Χάγης 1980 για τις απαγωγές των παιδιών. Ε, μπορείτε επιτέλους να θέσετε ένα τέλος σε αυτή τη διαμάχη, σε αυτή τη διαφωνία και να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αρμοδιότητα σε διεθνείς περιπτώσεις απαγωγής παιδιών. Ευχαριστώ. Ζωάλ Μπερσερών από το EFTD για 1,5 λεπτό. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Επομένως, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ε, Επιτροπής Γιούρι, δεν υπάρχουν άλλα μέλη της Επιτροπής Γιούρι που θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Δίνω το λόγο στην κυρία Ράιχερτς. Από ό,τι φαίνεται παίρνουμε πλέον το λόγο εμείς από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων για τις Γυναίκες. Και ε, με την παρουσία τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών εδώ, εμείς ήμασταν οι τελευταίες που έχουμε τη δυνατότητα τώρα να θέσουμε ερωτήσεις και ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα αλλάξει αυτή η διάταξη. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινούμε με τις ερωτήσεις των συντονιστριών από την ε, πλευρά της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις Γυναίκες. Εξ του ΕΛΚ, η κυρία Λεγκρίπ έχει το λόγο. Ένα λεπτό για να κάνει παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Ράιχερτς, θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στα θέματα των μισθολογικών ανισοτήτων. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2013 έκανε μια αξιολόγηση και είπε ότι η οδηγία σε σχέση με την ε, ισότητα ευκαιριών και ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα θέματα εργασίας δεν είναι επιτυχημένη, η οδηγία δεν εφαρμόστηκε σωστά και δεν μείωσε το χάσμα ε, των μισθολογικών ανισοτήτων που βασίζονται στο φύλλο. Ποιες είναι οι προτάσεις σας ποιες είναι οι θέσεις που θα υπερασπιστείτε, έστω και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που θα ασκήσετε τα καθήκοντά σας. Το Μάρτιο του 2013 εκδόθησαν ε, συστάσεις όχι το Μάρτιο 2014 διορθώνω, εκδόθησαν ε, συστάσεις. Είναι αρκετές ε, για να μπορέσετε να δουλέψετε σε αυτούς τους τέσσερις μήνες που θα ασκήσετε τα καθήκοντά σας. Και επίσης, τι ακριβώς σημαίνει ε, εργασία ίσης αξίας. Δεν έχει οριστεί αυτό με σαφήνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να πετύχουμε ε, ε, και πρόοδο. Άλλωστε έχουμε μια εσωτερική αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων. Ε, ρωτώ λοιπόν για τις μισθολογικές ανισότητες και να μιλήσω και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχετε προτάσεις για να προωθήσετε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, thank you, Κυρία Λεγκρίπ, σας ευχαριστούμε η κυρία Αρέν από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Όντω είναι δύσκολη άσκηση η σημερινή, διότι πρέπει να ε, δικαιολογηθείτε για το παρελθόν και ενδεχομένω να δεσμευτείτε για το μέλλον. Θα ήθελα τώρα, όπω και οι συνάδελφό μου, να σα ρωτήσω για τη θέση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Δεν είναι επαναλαμβάνω. Η δεύτερη σχετίζεται με την άδεια μητρότητα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μια πρόταση οδηγίας για μια καλύτερη προστασία των γυναικών ε, που εγκυμονούν ε, ή που θυλάζουν ε, και ο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αυξηθεί το ποσοστό αποσχολησιμοτητα ε, των γυναικών ε, και ε, η πρόθεση να καταργήσει αυτή την οδηγία αντιβαίνει σε αυτό το στόχο. Το αντίθετο, χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία οι γυναίκε όταν βρίσκονται σε αυτή τη θέση και εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε διεκπαιρεώσει σημαντικότατο έργο σε αυτό το τομέα. Απλή ερώτηση λοιπόν, δεσμεύεστε να συνεχίσετε αυτό το έργο και κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας η συγγήτρια, η κυρία Μωρέτη, που είναι Ιταλίδα, έχει αναλάβει ήδη τη δέσμευση να συνεχίσει τον αγώνα για αυτό το ζήτημα. Σα ζητούμε να ε, συνεχίσετε λοιπόν το έργο που έχει ήδη υλοποιηθεί και έχει να αρχίσετε από το μηδέν και πάλι. Ευχαριστούμε. Από πλευρά των φιλελευθέρων, η κυρία Λίναρ. Ευχαριστώ. Ε, καλωσορίσατε. Θα ήθελα ε, να αναφερθώ στην έκθεση Παρβάνοβα ε, που εγκρίθηκε στο τέλος της προηγούμενης ε, θητείας. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μία έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, το Φεβρουάριο του 2014 ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μία νομοθετική πράξη θεσπίζοντας μέτρα για την προώθηση της δράσης ε, στο πλαίσιο ε, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Πρόσφατα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραθέτω ότι δεν κρίνει πρόσφορο να υποβάλει νομοθετική πρόταση για προληπτικά μέτρα τέλος της παράθεσης. Ε, είναι πολύ απογοητευτικό διότι η έκθεση δεν ζητούσε υπερβολικά ε, νέα μέτρα. Σας απευθύνω απευθείας στην ερώτηση λοιπόν. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση που λάβαμε ως απάντηση. Και δεύτερον, τι προτείνετε να κάνετε για να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από νομοθετικής πλευράς. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που θέσατε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα εξ ονόματος της ECR θα λάβει τον λόγο η κυρία Φων Στόρχ. Παρακαλώ. Σα Dank. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Ράχερτ, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΩΣΑ ή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν τη συνεισφορά από πλευράς εργασίας και την οικονομική συνεργα... Ε, το οικονομικό έργο των γυναικών όσον αφορά τις μητέρες ε, που 24 ώρες ε, το 24ωρο εργάζονται και χωρίς ε, δικαίωμα διακοπών και έχουμε εδώ και θέματα συνδικαλιστριών, συνδικαλιστών και της μέρημνας των παιδιών. Σε σχέση με την ενισχύ τη διάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συνεισφορά των γυναικών από πλευράς εργασίας αναγνωρίζεται μόνο αν έχουν σύμβαση απασχόλησης και εργασίας οι γυναίκες. Τότε θεωρούν ότι είναι παραγωγή ε, για την κοινωνία. Αν έχουν όμως παιδιά και ασχολούνται με την ανατροφή τους, ε, τότε δεν θεωρείται ότι είναι παραγωγικό το έργο. Και τι θα γίνει σε σχέση με την μέρημνα και την ε, προσπάθεια ανατροφής των παιδιών. Θα είναι λιγότερο χρήσιμη. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστούμε. Και τώρα εξ ονόματος της ΓΚΟΕ Ενωτικής Αριστεράς η κυρία Μπιόρκ παρακαλώ. Thank you. ευχαριστώ. Πολλά θέματα είναι σημαντικά όπως η βία κατά των γυναικών, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, οι γονικές άδειες, η γονική άδεια για τις γυναίκες. Είναι στεναρή άποψή μας ότι η οικονομική και κοινωνική διάσταση από πλευράς των δικαιωμάτων των γυναικών δεν διασφαλίζονται επαρκώς και είναι οι πιο ηλικιωμένε γυναίκες εκείνες που βρίσκονται ε, ε, στα νοικοκυριά τους ε, και η ανάγκη περίθαψης που είναι δεδομένη δεδομένοι είναι περιορισμοί. Η ισότητα των φύλων πρέπει να μας κάνει να αυξήσουμε την ανεξαρτησία των γυναικών. Αυτό είναι στόχος μας, αλλά δεν υπάρχει δράση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και είναι συλλογικό σώμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά των Επιτρόπων. Είσαστε, έχετε την προθυμία να αναλάβετε λοιπόν κάποιες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της ισότητας των γυναικών. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα και κάποιος πρέπει να υπομειστεί τις ευθύνες. Τι θα κάνετε ώστε να υπάρξει ίση ανεξαρτησία από πλευρά των γυναικών και ιδιαίτερα για τις ηλικιωμένε γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα εξ ονόματος ε, των Πρασίνων, ο κύριος ε, Γιώργη Σεμπαστιά παρακαλώ έχει τον λόγο. Κυρία Ράχετσες τις επόμενες εβδομάδες η Ισπανική κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα μέτρο για τις εκτρώσεις ε, που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Η κατάσταση θα είναι ίδια όπως πριν από 20 ή 30 χρόνια ε, στο παρελθόν. Πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την κατάσταση. Ποια θα είναι η δράση που θα αναλάβετε σε σχέση με αυτή την οπισθοδρόμηση που θα είναι τρομερή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης για το ότι τηρήσατε τον χρόνο και Τέλος θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος ε, της, ε, ε, κυρία Αγιούτο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Ράιχετς. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ. Η Ιταλία έχει ένα πολύ χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στις, στην αγορά εργασίας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο μεταξύ των ηλικιών 15 ετών και 29 ετών υπάρχει μια κρίσιμη κατάσταση για την απασχόληση ιδιαίτερα των ε, νερών μητέρων και διαπιστώνεται ότι η κατάσταση των νερών μητέρων στην Ιταλία έχει επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ε. Και προφανώς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα έχουν το δικαίωμα να καταλήγουν και να έχουν πρόσβαση σε μια εξωτερική απασχόληση. Τότε θα πρέπει να έχουν και δυνατότητες όμως ε, παιδικών σταθμών, ε, ε, νηπιαγωγείων για τα παιδιά τους. Τι θα κάνετε λοιπόν ώστε τέτοιου είδους δημόσιες υπηρεσίες να διασφαλίζονται για αυτές οι γυναίκες και η διαθεσιμότητα να διασφαλίζεται για τα παιδιά τα οποία ζουν στο νότο της Ιταλίας. Τι θα κάνετε υπέρ αυτών. Πώς θα ενθαρρύνετε τις τοπικές αρχές να εφαρμόζουν και να υλοποιούν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τα νήπια, για τα μικρά παιδιά. Ποια μέτρα θα αναλάβει και διαβήματα θα, σε ποια διαβήματα θα προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τέτοιου είδους υπηρεσίες να διασφαλίζονται ιδιαίτερα για τους, ε, πιο μειονεκτικ... τους ε, ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε τον χρόνο και τώρα η κυρία Έχετε θα τον λόγο για να απαντήσει στι παρεμβάσει και ερωτήσει από πλευρά και των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών προηγούμενα. Ευχαριστώ. Voilà, euh, Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις τόσο συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις. Ε, τομείς που ενδιαφέρουν τους πολίτες, ε, τις γυναίκες, τους άντρες. Ε, πρόκειται για θεμελιώδη ερωτήματα. Θα αρχίσω με το εμπορικό δίκαιο και την αφαιρεγγιότητα. Έχουμε καλά νέα. Προς το παρόν υπήρξε μία σύγκληση απόψεων στο Συμβούλιο για το Συντονισμό Διαδικασιών που εκκινούνται σε περίπτωση αφαιρεγγιότητα στο Συμβούλιο. Οι τροπολογίες που κατέθεσε το Κοινοβούλιο εγκρίθηκαν Έχουμε αρχίσει τις επαφές ε, με το Συμβούλιο για να προχωρήσουμε την περαιτέρω προς την κατεύθυνση που ορίσατε. Για το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του τρέχοντος πιστεύω μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Εδώ λοιπόν ένα φάκελο στον οποίο θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Για τα δημόσια έγγραφα τώρα άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα για τους πολίτες ε, και η κατάργηση του web tape, δεν ξέρω πώς το λένε στα γαλλικά, δεν πειράζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα κείμενο σε σχέση με τη μείωση ε, των τυπικών διαδικασιών για την πρόσβαση ε, στα δημόσια έγγραφα και την ε, περαιτέρω διάθεση σημαντικών δημοσίων εγγράφων ε, Ορισμένε φορέ σε τέτοια <coughs> ζητήματα όταν έχουμε υπερβολικέ φιλοδοξίε δεν πετυχαίνουμε τελικά τίποτα και ε, πιστεύω ότι σχετικά γρήγορα μπορούμε να έχουμε μια ε, ικανοποιητική πλειοψηφία στο Συμβούλιο αν δεν είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Για την, τα έγγραφα της προσωπικής κατάστασης ε, ή της οικογενειακής κατάστασης νομίζω αυτό ε, παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους πολίτες. Λοιπόν, πιστεύω ότι συντομότατα μπορούμε να καταθέσουμε νέες προτάσεις διότι ξαναλέω στην Ευρώπη του σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το ζήτημα. Η Ιταλική Προεδρία τώρα. Είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί τη ε, και επιθυμεί επίση να προωθήσει αυτό το ζήτημα. Είμαι σίγουρη ότι στη δεύτερη ανάγνωση θα καταλήξουμε σε συμφωνία και θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για να καλύψουμε τις ε, πραγματικές ε, ανησυχίες των πολιτών. Το θέμα τώρα των γυναικών στα διευθυντικά συμβούλια είναι ένα θέμα κοινής αρμοδιότητας των δύο επιτροπών. Σας ευχαριστώ που θέσατε το ζήτημα. Όντως, η κυρία Ρέντινγκ ε, έκανε πολύ σημαντικό έργο σε αυτό το τομέα και είστε όλοι μάρτυρες ε, των ε, αγώνων που έγιναν σε αυτό το τομέα και εδώ ε, προτίθεται η Ιταλική Προεδρία να προωθήσει αυτό το ζήτημα. Έχει θέσει δε και ένα ξεκάθαρο στόχο να καταλήξει σε συμφωνία ε, πρωτού Οπότε σε αυτή τη σύντομη θητεία μου θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθήσω αυτό το σημαντικό φάκελο. Για την εξαίρεση για τις ε, επιχειρήσεις που υποεκπροσωπείται το γυναικείο φύλλο λιγότερο από 10% του εργατικού δυναμικού η ιδέα ήταν να δείξουμε ευελιξία πιστεύω όμως ότι μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία του Κοινοβουλίου για την κατάργηση αυτής της εξαίρεσης ως προς τις κυρώσεις θα υποστηρίξω την ε, τροπολογία για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, ε οι προτάσεις ενίσχυσης μου φαίνονται δυσανάλογα φιλόδοξης. Μπορούμε νομίζω να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα. Κανονισμός Βρυξέλλες 1. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποιος ε, έκανε την ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη. Μπερδεύτηκα λίγο. Λοιπόν, Βρυξέλλες 1. Στην ε, μεταρρύθμιση ε, το σημαντικό στοιχείο είναι η κατάργηση του εκτελεστού τίτλου. Νομίζω αυτό είναι ε, το σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να καλύψει τις διεθνείς πτυχές. Δυστυχώς πλειοψηφία στο Συμβούλιο αυτό το ζήτημα δεν ευρέθη. Στι Βρυξέλλες 1 υπάρχει ρήτρα αναθεώρηση και οι νομικές μας υπηρεσίες ήδη επεξεργάζονται αυτή ακριβώς τη διάταξη. Σας ε, ευχαριστώ ε, για την ερμηνεία που δίνετε τη δράση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, γιατί όντω ε, είναι ένα από τα χέρια σημασία θέματα για μας. Για το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων ξέρω είναι δύσκολο το ζήτημα και υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό μάλλον σχετίζεται ε, με το ότι ε, αυτό το ζήτημα ε, αποτελεί ουσιαστικά τον πυρήνα του αστικού δικαίου σε πολλά κράτη-μέλη. Κάποιοι θέλησαν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογή στι επιγραμμικές πωλήσει με την ελπίδα να τυχηθούν και άλλα, ναι, και άλλα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο στην πλειοψηφία που έχουμε ήδη. Θα παραμείνουμε σε επαφή και θα δούμε τις εξελίξεις. Υπάρχει και μία άλλη επίκριση που ακούμε συχνά ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, ε, περιορισμένη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σας θυμίζω ότι είναι προαιρετικό το σύστημα. Ο καταναλωτής πάντοτε έχει τη δυνατότητα, εξυπακούεται, να πάει να κάνει τα ψώνια του εκεί όπου θέλει. Ε, το κράτος δικαίου. Ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε, μιλήσαμε ε, πολύ για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα, πραγματικά είναι ακρογωνίως λίθος της δημοκρατίας και σωστά είπατε πως ανέκυψαν διάφορα προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία για το κράτος δικαίου να υποβάλει μια ανακοίνωση. Το άρθρο 7 είναι η πυρηνική βόμβα, όπως λέει ο πρόεδρο Μπαρόζο και η ανέκαθεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ακολουθούσε αυτή την προσέγγιση του πικοδομητικού διαλόγου με τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης ε, ενώ ανάμεσα στα κράτη-μέλη υπέβαλε αυτή την ανακοίνωση περιγράφοντας τη διαδικασία που έχει ήδη ακολουθήσει και προτίθεται να ακολουθήσει σε περίπτωση που ε, προκύψει και πάλι τέτοιο ζήτημα. Αμοιβή αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων σε θέματα αστικού δικαίου και αναφερθήκαμε σε αυτό και ε, πώς δηλαδή στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε μια καλύτερη γνώση των πολιτών για τα δικαιώματά τους που κατοχυρώνται ε, ε, στο δίκαιο. Νομίζω ότι αυτό το έργο μπορώ να το συνεχίσω, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε παραδείγματο χάρη τα δικαιώματα ε, των ε, μερών ε, θεσπίζοντας ελάχιστα κριτήρια Αναφερθήκατε επίσης στη δικτυακή πύλη e-Justice. Εσείς μου κάνατε την ερώτηση. Όλα αυτά ε, τα εργαλεία μας επιτρέπουν ε, να έχουμε μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσματικότερες δράσεις για την ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου. Ο πίνακας επιδόσεων, αναφερθήκατε και σε αυτό, όντως είναι ένα ζήτημα διαφάνειας. Πρέπει να δούμε σε ποιο στάδιο έχει γίνει η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Κύριε Καβαντά, μου μιλήσατε για τις... Ε, για τα γαμικά καθεστώτα και ε, δεδομένης της κατάστασης και της μετεξέλιξης των ε, ηθών ε, νομίζω ότι όντως θα πρέπει να ασχοληθούμε εντατικά με αυτό το ζήτημα όμως θα πρέπει να διασυνδεθούν αυτά τα δύο ζητήματα της κληρονομικής διαδοχής δηλαδή και των γαμικών καθεστώτων για να υπάρχει μια ακολουθία και οι δύο πτυχές θα πρέπει από κοινού να εγκριθούν από τα πλευράς τακτικής νομίζω ε, είναι σημαντικό να ε, ε, παραμείνουν διασυνδεδεμένα αυτά τα ζητήματα στο τρίο της Προεδρίας όπως είναι γνωστά, γνωστό στα γαλλικά ακούγεται περίεργο τέλος πάντων αυτή η άτιμη δομή σε συνδυασμό με την Ιταλική Προεδρία μας προσφέρουν εχέγγυα για να άρουμε τα τελευταία κολλήματα και σας θυμίζω ότι χρειαζόμαστε ομοφωνία για αυτό το θέμα. Ε, από τεχνικής πλευράς λοιπόν συνεχίζονται οι διαδικασίες και πιστεύω ότι προχωρούμε. Η οθεσία παιδιών ε, νομίζω ότι ε, το ζήτημα αυτό δεν ρυθμίζεται σε κάποιο νομοθέτημα. Κινούμεθα στα πλαίσια της Σύμβασης της Χάγης, όπως το θυμήσατε. Υπάρχει το θέμα της ε, αμοιβαία αναγνώρισης ε, των διαδικασιών υιοθεσία. Κύριε Καβαντά, εσείς αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα, αν δεν κάνω λάθος, με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την κατάσταση να έχει υιοθετηθεί ένα παιδί σε μία χώρα και σε μία άλλη να μην αναγνωρίζεται η υιοθεσία. Έχουμε πλήρη επίγνωση του προβλήματος, γιατί και πάλι πρόκειται για θέματα της καθημερινότητάς μας. Ε, κάναμε μία μελέτη, δεν θέλω να ακούγομαι και πολύ γραφειοκρατική, τέλος πάντων. Κάναμε μία μελέτη και τελικά ε, ε, σκοπεύουμε να λάβουμε πρωτοβουλία τους ώστε να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση των πράξεων ε, οικογενειακής κατάστασης. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα έχει κέρια σημασία. Θα ζητήσω από το Συμβούλιο να επιταχυνθούν οι εργασίες ε, διότι ε, μπορούμε να ρυθμίσουμε, όχι με όμορφο τρόπο, αλλά μπορούμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των πράξεων οικογενειακής κατάστασης. Λοιπόν, για τις απολαυές των γυναικών ε, στρέφομαι τώρα ε, στις ερωτήσεις της Επιτροπής Γυναικών. Όντως ε, υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Γυναίκα είμαι και εγώ, δεν πρόκειται να το διαψεύσω. Νομίζω προς το παρόν είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με τα θέματα διαφάνειας. εγώ πιστεύω πολύ στη δύναμη της peer pressure, της πίεσης από πλευράς των ομολόγων και ομοτήμων μάλλον τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ακολουθήσουν τις ε, συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γραπτό το 2015 να μας κοινοποιήσουν ε, τα αποτελέσματα των μελετών που θα κάνουν για να εξεταστεί η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Ε, για τη βία κατά των γυναικών και πάλι εδώ ε, Ω θεματοφύλακα των συνθηκών, η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα ε, για αυτό το ζήτημα. Δεν μιλήσαμε πολύ για τη διαδικασία σε παραβάση, αλλά όταν συντρέχουν οι νομικέ προποθέσει, αλλά αυτό είναι θέμα εφαρμοστέου δικαίου, όντω είναι σημαντικό να κινούνται οι διαδικασίε. Πρέπει να προτείνουμε μια οδηγία για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών. Ξέρω, ξέρω ότι η κυρία Κασιά Πέρες ε, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα και η Επιτροπή της φυσικά. Υπάρχει το πλαίσιο ελέγχου σίγουρα, αλλά από πλευρά ποινικού δικαίου για την ανάληψη πρωτοβουλίας ε, θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού το θέμα της νομικής βάσης, διότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι και προς το παρόν θεωρούμε ότι είναι κάπως δύσκολο. Ε, υπολογίζω στην ευρηματικότητα της Επιτροπής ε, ε, Γυναικών, κύριε Γκασία Πέρες, για να βρεθούν ε, καινοτόμες λύσεις. Ε, άδεια μητρότητας. Εδώ και πάλι σχολιάζεται το ζήτημα ο υποψήφιος πρόεδρος Γιούνκερ ε, σχολίασε το ζήτημα. Νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί πολλά για αυτό το θέμα. Η οδηγία εδώ και χρόνια ε, είναι πάνω στο τραπέζι και με κάπως μηχανικό τρόπο ε, έχουμε ε, ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία η οποία έχει καταλήξει ένα τέλμα. Δεν έχει συμβεί τίποτα ε, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, η Ιταλική Προεδρία φιλόδοξη αποφάσισε να ανακοινήσει το ζήτημα και ξαναλέω γυναίκα είμαι, δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία. Και μπορώ να πω ότι αυτή η πρώτη οδηγία, αν αποφασίσει να κινηθεί το Συμβούλιο και έτσι φαίνεται, θα ακολουθήσει τη συνήθεια εδώ. Σημαντικό είναι να συνδράμουμε την Ιταλική Προεδρία και τα κράτη-μέλη σε αυτή τη νέα προσπάθεια που θα κάνουν. Ήδου, Πρόεδρε, ε, πιστεύω ότι όντως έκανα ε, το γύρο, απάντησα σε ερωτήσεις, σίγουρα ε, πολύ γρήγορα, αλλά πιστεύω ότι απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις που με έθεσαν τα μέλη των Επιτροπών. Σα ευχαριστώ. Θα σας ρωτούσα κυρία Ράχερτς, αν μπορείτε να απαντήσετε συντομία τις ερωτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όμως, αυτά τα οποία είπατε νομίζω ότι δείχνουν ότι ε, και οι τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, θεωρούν ότι δώσατε πολύ περιεκτικές απαντήσεις, πολύ ολοκληρωμένες για μια προσωρινή θέση. Άλλωστε, έχετε περάσει από μια πλήρη ακρόαση κοινοβουλευτική ενώ ε, θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας για τέσσερις μόνο ε, μήνες. Θεωρώ ότι δεν θέλετε να κάνετε καμία ε, καταληκτική δήλωση. Θέλουμε μόνο να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσουμε τους συντονιστές από τις τρεις κοινοβουλευτικέ επιτροπές, να ευχαριστήσουμε και τα μέλη που είναι εδώ στην αίθουσα, γιατί είναι μια κατεξαίρεση διαδικασία δεν θα γίνει η ίδια διαδικασία με τις υποψηφιότητες των νέων επιτρόπων. Ε, εκεί θα έχουμε μια πλήρη ακρόαση με πάρα πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ όλους να ζητήσω από τους συντονιστές μόνο να παραμείνουν στην αίθουσα για να κάνουμε την αξιολόγηση της κυρίας Ράχερτς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ράχερτς και όλους τους υπόλοιπους.